σημείο αυτό μέτρα και αυτό θα σημαίνει αλληλεγγύη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, με τους δημόσιους οργανισμούς. Ευχαριστούμε κύριε Μαν. Πριν περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye, μου έχει κατατεθεί μια ανακοίνωση που θέλω να σας τη διαβάσω. Δηλαδή οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας ανακοίνωσαν ότι ο κύριος Σίας Ντερόσα από τις 15 ε, Φεβρουαρίου του 2012 ε, θα αντικατσαθεί από την κυρία Κοστέλο και εγώ ε, καλωσορίζω την ναι, δεν ξέρω, ήρθε ήδη, εδώ είναι. Γεια σας, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού του Κοινοβουλίου όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρίες του Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα όσο η ε, θητεία τους ε, δεν αμφισβητείται και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μέλος ε, δήλωσε γραπτά ότι δεν κατέχει άλλη θέση που να αντιβαίνει, να μη συμβαδίζει με την θέση της Ευρωβουλευτού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Και τώρα πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, έχω λοιπόν την εξής κατάσταση μπροστά μου.